αρχίσουμε σε αυτόν τον τόνο τις προσωπικές τοποθετήσεις. Την Τετάρτη θα προσυπογράψουμε 22 αποφάσεις ε, συναπόφασης βάσει και του άρθρου 74 του κανονισμού και στις 15 του μήνα θα έχουμε και την υπογραφή για τον δημοσιονομικό κανονισμό. Και όλα αυτά βάσει της ε, χθεσινής μας συζήτησης και των πρακτικών από τη χθεσινή σύνοδο. Ας περάσουμε λοιπόν στην ημερήσια διάταξη. Το επόμενο σημείο προβλέπει την δήλωση του διορισμένου Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στον Ζωζέ Μανουέλ Μπαρόζο.